Ευρωπαϊκή Ένωσης να θίξει το θέμα στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα γίνει με την Ινδία στα τέλη Ιανουαρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεχούιχτ. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν έξι ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί από τους πράσινους, την ΚΟΕ, το ΕΛΚ, τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές, τους συνδυατικούς και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της συζήτησης. Το επόμενο θέμα αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν. Ο κύριος Σλίτερ για ένα λεπτό από του συντάκτες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια είπαμε ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν έριξε αέρια ε, σε ειρηνικούς διαδηλωτές. Είδαμε τα βασανιστήρια, ε, τη φυλάκιση, την απαγόρευση ταξιδιών. Ένα έχω μόνο να πω στις αρχές του Μπαχρέιν, σταματήστε επιτέλους. Μέσα στο ψήφισμά μας ε, βλέπουμε την απαγόρευση, τα διάφορα μέσα καταπίεσης ε, που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση του Μπαχρέιν πέρα από τα αέρια ε, που ρίχνει στους διαδηλωτές και την απαγόρευση ταξιδιών. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ΙΕ πρέπει να δράσει για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές προτού αρχίσει ο εμφύλιος στο Μπαχρέιν ε, και το ίδιο ισχύει για τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα σκέφτομαι έναν ε, Σουηδό Μοχάμετ Αλμουάτ που είναι στην φυλακή στον Μπαχρέν και για τους οποίους δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλούτερ. Ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω σαφές ότι πολλά από αυτά τα οποία έχουν λάβει χώρα στην, στο βασίλειο του Μπαχρέν μετά από τις αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες είναι απαράδεκτα η αστυνομία έχει δράσει με δυσανάλογη βία και πολλοί διαδηλωτέ έχουν σκοτωθεί. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτέ τι ακρότητε και αυτά τα εγκλήματα πρέπει να έρθουν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Η ομάδα μου, η συντηρητική, συμμερίζεται την ανησυχία όλων ομάδων για το γεγονό ότι έχει αφαιρεθεί και η ηθαγένεια πολλών από του διαμαρτυρόμενου και επίση φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα για την ελευθερία έκφραση και την αμεροληψία τη δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι υπαρξιακέ απειλές προς το βασίλειο του Μπαχρέιν που προέρχονται ιδίω από το Ιράν. Οι προσπάθειες του Ιράν να ε, ανατρέψει την κυβέρνηση αν επιτύχουν θα είναι πραγματικά ε, ολέθριες. Ενώ πρέπει να υπάρξει μια διερεύνηση για όλα τα θέματα αυτά που αναφέραμε, όλοι θέλουν να υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή στον Μπαχρέν, η οποία να ενδεσμευμένη για όλους, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ακολουθεί κυρία Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μπαχρέιν είναι μία από τις αραβικές χώρες όπου η αραβική άνοιξη οδήγησε σε μία γενικότερη λαϊκή κινητοποίηση, η οποία κατεστάλλει με βία. Αυτή η καταστολή έγινε με τη βοήθεια του στρατού της Σαουδικής Αραβίας που γνωρίζουμε πολύ καλά το ρόλο τους εδώ και δύο χρόνια. Η καταστολή δεν έχει σταματήσει, οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων συνεχίζονται και πολλαπλασιάζονται. Θέλουν να μας δώσουν την εντύπωση ότι είναι μια εθνικό ε, θρησκευτική σύγκρουση μεταξύ μια μειονότητα Σουνιτών και μια πλειοψηφία Σιητών. Αλλά όπω και στην Τινησία πρόκειται πάνω απ' όλα για οικονομικέ και κοινωνικέ διεκδικησει διεκδικήσεις. Αλλά πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν διακόψει τι οικονομικέ του σχέσει με τον Μπαχρέν και ιδίω δίνοντας όπλα και εργαλεία για την καταστολή όπως είναι το τα δακρυγόνα και μέσα για, την, για τον έλεγχο των διαδηλωτών. Τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει επιτέλους αυτές τις εξαγωγές. Θα είναι τουλάχιστον ένα δείγμα κύριε Επίτροπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρθεί στο ύψος του βραβείου Νόμπελ της Ειρήνης που έχει λάβει. Ευχαριστώ. Κυρία Βεζιά. Ακολουθεί η κυρία Ευχαριστώ. Ως ε, μέλος της Επιτροπής ε, της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το θέμα αυτό, επισκέφθηκα τον Μπαχρέιν πριν από ένα μήνα. Ελπίζουμε ο πολιτικός διάλογος και η οικονομική συνεργασία να αναπτυχθούν περαιτέρω επί της σωστής βάσεως. Ωστόσο, δεν μπορούμε και δεν θα αγνοήσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες ε, ε, ε της ε, ε, περιοχής και στο Μπαχρέιν πιο συγκεκριμένα. Κρατήθηκαν στη φυλακή 13 επιφανείς ακτιβιστές ε, με την κατηγορία ότι ε, προσπαθούν να χτυπήσουν τη μοναρχία. Η πιο γνωστή είναι ο κύριος Ιμπραχήρ Σαρίφ, ε, είναι από τους φυλακισμένους τους οποίους επισκεφθήκαμε όταν πήγαμε στο Μπαχρέν και έχουν καταστεδαστεί σε ισόβια ποινή και μόνο μια δημόσια χάρη θα αλλάξει τη μοίρα τους. Κάνω έκκληση να ε, απελευθερωθούν όλοι οι ε, κρατούμενοι λόγω συνειδήσεως και να ξεκινήσει ένας ε, εντατικός εθνικός διάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Αντρικάινε. Η κυρία Ούλαντια δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως τμήμα της Αραβικής Άνοιξης, οι διαμαρτυρίες στο Μπαχρέιν ως στόχο είχαν να επιτύχουν περισσότερη πολιτική ελευθερία και ισότητα για τον ε, πληθυσμό των ζητών, ε, ε, αλλά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δυστυχώς η εξουσία δεν έχει επιτρέψει ακόμα να ξεκινήσει μια ελεύθερη συζήτηση επί του θέματος αυτός και αντί να έρθει σε επαφή με τους ε, διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας ε, κατέστηλαν αυτές τις διαδηλώσεις. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες δυστυχώς το Κοινοβούλιο ε, παραβίασε τα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων στην ελεύθερη διαδήλωση, στο ελεύθερο ραδιόφωνο και στην ελευθερία του λόγου. Επιπλέον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως και κάποια θετικά στοιχεία κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ο διορισμός ενός ε, ombudsman. Ε, το ψήφισμα αυτό δεν έχει στόχο να παρέμβει στα εσωτερικά ζητήματα του Μπαχρέιν. Επικεντρώνεται στην ανάγκη να σεβαστούμε τις ε, δημοκρατικές αξίες και να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Χωρίς ε, διάλογο μεταξύ των σιτών που είναι η πλειοψηφία του Μπαχρέιν, η κυβέρνηση ε, απομακρύνεται από τη δημοκρατία. Και ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να σταματήσει να καταστέλει όλες τις διαδηλώσεις και να απελευθερήσει όλους τους φυλακισμένους ακτιβιτές και να βοηθεί, ε, επιτρέψει να ε, ε, υπάρξουν οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Ακολουθεί ο κύριος Ρέπο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς η κατάσταση στον Παχρέν έχει παραμείνει αναλύωτη. Από τον προηγούμενο Δεκέμβριο γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες, έχουμε βρεθεί στον Παχρέν, έχουμε μιλήσει με πολιτικούς κρατούμενους, αλλά η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ σοβαρή. Πρέπει να κατανοήσουμε συγχρόνως ποιο είναι το γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται εκεί το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του δίνει ένα μήνυμα καλής θέλησης. Συγχρόνως εμείς απαιτούμε οι υπεσχημένε μεταρρυθμίσεις να λάβουν χώρα πράγματι και να υλοποιηθούν. Το καθεστώς του Μπαχρέιν θα πρέπει να προχωρήσει σε πραγματικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες του Μπαχρέιν έχουν κατέβει στον δρόμο ζητώντας να γίνουν ακουστές οι απόψει του και τα αιτήματά του και να έχουμε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κάτι μελη θα πρέπει να πράξουν το ότι μπορούν καλύτερο για να του βοηθήσουν ώστε να υπάρξει ελευθερία στο Μπαχρέν. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο, οι ομιλητέ των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Βάιντερ, πρώτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το Δεκέμβριο του Δεκεμβρίου εγώ πήγα με την αντιπροσωπεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και είδαμε την κατάσταση που επικρατεί με τον αγώνα εναντίον μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό ήδη σε επίπεδο υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γι' αυτό εκπλήσωμε, γιατί το θέμα αυτό παρουσιάζεται ως θέμα κατεπήγοντος. Προφανώς υπάρχει ένα υπόβαθρο που είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων που δεν βασίζονται σε δικαιακά στοιχεία σε σχέση με τους αντιπολιτευόμενους. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, έχουν γίνει αλλαγές στο Σύνταγμα του Μπαχρέιν, έχουν γίνει προσπάθειες να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας στην ε, αστυνομία Υπήρξαν λοιπόν πολλές προσπάθειες για να δοθούν απαντήσεις στα θέματα αυτά. Είχαμε πάντως τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους πολιτικούς κρατουμένους στις φυλακέ. Ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε σε μια μονομερή στάση και θα υποστηρίξουμε τον Μπαχρέιν. Κύριε Γκουρμά, για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Παρότι υπήρξαν κάποιε θετικέ εξελίξει στην αλλαγή τη χιλιετία, διότι μπορούν πλέον να ψηφίσουν, παραδείγματο χάρη οι γυναίκε, ε, άρχισε τα τελευταία χρόνια να επιδεινώνεται η κατάσταση στον Μπαχρέν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κρατικέ αρχέ κάνουν βασανιστήρια, ασκούν υπερβολική βία κατά των ειρηνικών διαδηλωτών και των ακτιβιστών ε, για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεθνεί οργανώσει για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να στείλουν τα μέλη του για να παρατηρήσουν την κατάσταση απαγορεύεται από τις ε, αρχές. Ε, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να συναυθεί από πλευρά των αρχών του Μπαχρέιν η σύμβαση για τους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης ε, για, κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι απαραίτητο. Οι πολίτες του Μπαχρέιν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα με ειρηνικό τρόπο να εκφράζουν τις πολιτικές τους απόψει, είτε στις διαδηλώσεις που γίνονται είτε μέσα στα κοινωνικά τεχνολογικά μέσα. Ε, στη συνέχεια ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν και οι γυναίκες ε, να ενισχύουν το ρόλο τους ε, στη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκουρμαή. Προσπαθούν οι διερμηνείς, αλλά ξέρετε ότι ό,τι και να κάνουν κάποια στιγμή δεν προλαβαίνουν. Σας παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά για να μπορούν να σα παρακολουθήσουν. για ένα λεπτό. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα έγκλημα παράδεκτο για οποιαδήποτε χώρα και να μιλάμε. Δεν μπορούμε να είμαστε συγκαταβατικοί σε σχέση με τη δράση τέτοιων κυβερνήσεων. Ε, το Μπαχρέιν είναι από τις χώρες ε, όπου είναι γνωστές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταστολή στοχεύει τους χριστιανούς, ε, δολοφονίες, διακρίσεις είναι συχνά φαινόμενα και γίνονται δεκτά από τις αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει καταδίκασε ήδη επανειλημμένα ε, αυτή τη στάση των αρχών του Μπαχρέιν, αλλά δεν επαρκεί αυτό. Θα ήταν πιο σημαντικό να δράσουμε ούτω ώστε να ανακόψουμε αυτή τη δράση. Αφήστε που έχουμε και ένα ατού για να, ε, με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσουμε την κοινότητα των χριστιανών. Ευχαριστώ κύριε Γκρόμπαρτσέκ. Ακολουθεί ο κύριος Μέρφυ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δύο σχεδόν χρόνια ο λαός του Μπαχρέιν αντιμετωπίζει μια τεράστια καταστολή και επιθέσεις από μια κυβέρνηση που είναι διατεθειμένη να μην παραχωρήσει κανένα ουσιαστικό ανθρώπινο ή δημοκρατικό δικαίωμα. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν υπολογίζει ότι έχουν γίνει περίπου 100 εξοδικαστικές εκτελέσεις τα τελευταία δύο χρόνια και πάνω από 800 άτομα μεταξύ των οποίων και ανήλικοι έχουν μπει στη φυλακή επειδή διαμαρτυρήθηκαν και ιδίως οι συνδικαλιστές. Υπάρχουν επίσης απαγωγές, σεξουαλική βία και βασανιστήρια. Είναι πραγματική υποκρισία. Οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις να μιλάνε για την ανάγκη για δημοκρατία στην περιοχή από τη μία πλευρά, από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Βρετανία εξακολουθούν να δίνουν όπλα σε αυτό το καθεστώ, ιδίω δακρυγόνα τα οποία χρησιμοποιούνται και σε περιοχέ όπου δεν υπάρχουν διαδηλωτέ. Όλα τα συμβόλαια αυτά πρέπει να σταματήσουν. Θα πρέπει να φύγει το φύλλο εκεί των ΗΠΑ από το Μπαχρέν και η συνεργασία με μέσα στα πλαίσια τη σχέση με τι χώρε του Περσικού κόλπου πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι αγωνιστέ και οι συνδικαλιστέ των αγώνων να αλλάξουν την κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Μέρφυ, οι υπόλοιποι ομιλητέ και πρώτο ο κύριο Λιέζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα προ την κυβέρνηση του Μπαχρέιν και να τονίσουμε ότι οι συνταγματικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα τύχουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο δεν θα υποστηρίξουμε είναι η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταστολή κατά της αντιπολίτευσης και η χρήση πρόσχημάτων ώστε η χρησιμοποίηση της, του αγώνα κατά της τρομοκρατίας ως προσχήματος για την καταστολή. Όλες αυτές τις πρακτικές θα πρέπει να καταδικαστούν. Θα πρέπει να είμαστε επίσης προσεκτικοί να μην ενοχοποιήσουμε όλο τον πληθυσμό. Ευχαριστώ κύριε Λίσεκ. Για μπλε κάρτα ή για οφθαλμοσύλληψη. Μπλε κάρτα. Κύριε Ελίζα, δέχόσαστε μια μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Σόνικ, Σόνικ λέγομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο συνάδελφος γνωρίζει ότι η κατάσταση στις Αραβικέ χώρες τι οποίες συζητούμε είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι νομίζουμε. Εγώ επισκέφθηκα τον Μπαχρέιν και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που επιτρέπει να κατασκευάζονται εκκλησίες για χριστιανούς και μάλιστα πολλοί ε, ε πηγαίνουν στην εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Το γνωρίζω αυτό το οποίο μου είπατε και το είπα σαφώς. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των θετικών στοιχείων και των αλλαγών που πρέπει ε, να γίνουν και που ανακοινώνονται. Οι αλλαγέ που ανακοινώνονται είναι μεν δημοκρατικέ, αλλά θα πρέπει να καταδικάσουμε και πράξει οι οποίε αντιβαίνουν τι δεσμεύσει αυτέ, ιδίω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Σάρβαμα. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να μην διαθέτουμε όλες τις λεπτομέρειες ε, για την έκταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παχρέιν, αλλά θα πρέπει να εκφράσουμε τη μεγάλη μας ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει πλέον να επικεντρωθούμε διεθνώ στο να στηρίξουμε τα θετικά στοιχεία του ζητήματο. Είναι θετικό, για παράδειγμα, ότι ο βασιλιά και η κυβέρνησή του ε, ενέκριναν την ε, ε, ανεξάρτητη έρευνα τη Επιτροπή του Μπαχρέιν και θέλουμε από εκεί και πέρα αυτά να τα ακολουθήσουν και αλλαγέ πραγματικέ επιτόπου. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι οι παραβιάσει κατά παιδιών απλώς και μόνο διότι είναι επονίδιστες και θα πρέπει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν να δράσει οποιαδήποτε κατηστολή ε, από πλευράς του κράτους, ανεξάρτητα από το που γίνεται και ποιο ε, κρύβεται πίσω από αυτό, ε, είναι καταδικαστία. Και μάλιστα είναι πάντα καταδικασμένη στην αποτυχία. Δεν μπορούμε πλέον να αφήνουμε τους ανθρώπους στο σκοτάδι για το τι συμβαίνει στη χώρα τους. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αργά ή γρήγορα θα σταματήσουν. Ακολουθεί η διαδικασία η διαδικασια είναι πάρα πολλοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Εγώ θα περιοριστώ σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει το λόγο ακόμα. Κύριε Σύνδεσκα, έχω διαφο... προβλήματα με το όνομά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν πειράζει που δολοφονείτε το όνομά μου. Το καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να δώσει προσοχή σε όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων ένα, αντιμετωπίζουμε θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βία κατά των πολιτών τους που ζητούν με μεταρρυθμίσεις πολιτικού χαρακτήρα. Όπως φάνηκε και από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μπαχρέιν που έχει επιβεβαιώσει την, την ε, καταδίκη σε ισόβια δεσμά ηγετών διαδηλώσεων πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει να καταδικάσουμε λοιπόν όλες αυτές τις περιπτώσεις ατιμορρησίας των κρατικών αρχών που στρέφονται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα πρέπει να δράσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα επικρατήσουν και θα επερευθερωθούν οι ακτιβιστές. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίσλευκα, κυρία Μακχοβ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να μιλήσω για τη βία κατά των ανηλίκων στο Μπαχρέιν. Τον προηγούμενο μήνα 80 ανήλικοι μεταξύ 15 και 17 ετών φυλακίστηκαν σε σοφρονιστικά ιδρύματα στο Μπαχρέιν. Ο Μοχάμεντ Μουχαμά, 16 ετών από τη Σίδρα, συνελήφθη στο σπίτι στις αρχές Δεκεμβρίου και τον στείλαν στις φυλακές χωρίς να έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή ούτε με την οικογένειά του ούτε με κάποιο δικηγόρο. Μετά από μερικές μέρες τον στείλαν σε ένα διαφορετικό σοφρονιστικό κέντρο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και ποτέ δεν του απεικέρθη κατηγορία, κανείς δεν ξέρει γιατί τον συλλάβανε. Αυτό είναι μονάχα ένα παράδειγμα. Θέλω να ζητήσω από τις αρχές του Μπαχρέν να σταματήσουν τέτοιου είδους ε, δράσεις κατά των ανηλίκων. Πάρα πολλέ φορέ. αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι αυτοί οι ανήλικοι έχουν συμμετάσχει μαζί με πιο, μεγάλα, πιο ενήλικου, ενήλικους σε εκδηλώσει διαμαρτυρία. Το δικαστικό σύστημα στον είναι επίσης να λειτουργεί με τρόπο αμερόληπτο και να τιμωρεί τους ε, κακού. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή μετά την Αραβική Άνοιξη πήραν θάρρο οι πολίτες ε, του Μπαχρέιν και κατέβηκαν στους δρόμου για να υπερασπιστούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τις πρώτες ειρηνικές ε, διαδηλώσει. Ε, δυστυχώς δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα. Παραμένει η ίδια η στάση των αρχών. Τρομοκρατούν τους ανθρώπου, Μαζική καταστολή. Παρόλα αυτά έχει αναλευθεί επίσημη δέσμευση για να αρχίσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις ε, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκροτήθηκε μέχρι και ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνηση ε, των ε, αιματηρών αυτών επιθέσεων και επίσης αναμενόταν η εκτέλεση του σχετικού ψηφίματο του ΟΗΕ. Μόνο σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμε και μακροχρόνιε λύσει για να σταθεροποιηθεί ε, η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Σας ευχαριστούμε η κυρία Γκέρνγκερ Ότιγκερ. Η κυρία Μπασέσκου για να κλείσει αυτός ο γύρος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Μπαχρέιν ε, παραμένει ανησυχητική. Η απόφαση των ΟΤΑ του δικαστηρίου ε, σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ε, την ανικανότητα του δικαστικού συστήματος να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξίσου με ανησυχεί το ότι αγνοούνται τα δικαιώματα των παιδιών στο Μπαχρέιν ε, διότι θεωρούνται ως ενήλικες ε, στο δικαστικό σύστημα και έχουμε διάφορες ε, καταγγελίες βασανιστήριων κατά ανηλίκων. Γενικά το δικαστικό σύστημα και το σύστημα επιβολής του νόμου στον Παχρέν πρέπει να μεταρρυθμιστεί άρδιν διότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπασέσκου. Περατώνεται στη διαδικασία κάτσε διάη και θα ακούσουμε τελική παρέμβαση του Επιτρόπου Τεγκούχτε. Πρόεδρε, Αξιότιμοι βουλευτέ, ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσω τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου σε σχέση με το να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα για την Ένωση αυτή η χώρα είναι υψίστη ε, σημασία σε αυτό το ζήτημα για την ύπατη εκπρόσωπο και την υπηρεσία εξωτερική δράση, ε, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τη βία από οποιαδήποτε πλευρά. Αυτό είναι ο πυρήνας των δράσεών μα. Οι πολυάριθμες δηλώσει και οι επαφέ που είχαμε με τι αρχές ε, καταδεικνύουν τη δέσμευσή μα Το ίδιο και όταν συναντηθήκαμε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ε, σημαντικό ζήτημα, ενώ η διαδικασία εσωτερικής ε, συμφιλίωσης ε, θα πρέπει να τροχιοδρομηθεί σε κρατεότερες βάσεις. Εκφράσαμε την ανησυχία μας επίσημα σε σχέση με την διατήρηση των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των ακτιβιστών ε, υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δοθεί χάρη ε, σε αυτούς τους ακτιβιστές ε, που κρατούνται στον Παχρέιν σε σχέση με τα συλλαλητήρια του 2011. Ο διάδοχος του θρόνου στον Παχρέιν έκανε ένα πρώτο βήμα ανοίγματο προς την αντιπολίτευση η οποία ανταποκρίθηκε και θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να προλιάνουμε το έδαφος και να επιτύχουμε μια πιο βιώσιμη λύση, να δράξουμε την ευκαιρία επίσης έτσι ώστε και πάλι να απευθύνουμε έκκληση προς αρχές του Μπαχρέου ε, για να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής Μπασέιν όπως ονομάζεται. Ε, στη συνέχεια έχουμε την καθολική αναθεώρηση για την κατάσταση στο Μπαχρέιν ε, που αναμένει στα τέλη του έτους θα δούμε ποιες θα είναι οι συστάσεις. Αυτό επίσης που χρειαζόμαστε είναι διάλογος με την κοινωνία των πολιτών για να ρυθμιστούν μακροχρόνια τα εκκρεμή ζητήματα. Καλούμε τις αρχές του Μπαχρέιν ε, να ασχοληθούν με τα αιτήματα των πολιτών για την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Ε, χρειάζεται εσωτερική συμφιλίωση, η οποία όμως ε, θα επιτευχθεί μόνο με παροχή εξωτερικής βοήθειας και τεχνογνωσίας. Τέλος, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την επίσκεψη τη αντιπροσωπεία στο Μπαχρέιν το Δεκέμβριο του 2012 θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου διότι είναι ιδιαίτερα ισορροπημένε και ορθολογικέ οι υπό επιτροπής. Σα ευχαριστούμε κύριε Τεκούχτ. Ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση για αυτό το θέμα. Έξι ψηφίσματα από του πρασίνου συντηρητικού, την Κούτσφελ Ελεύθερου, το ΕΛΚΑ και του σοσιαλιστέ έχουν